για τις αποζημιώσεις για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών και η παροχή βοήθεια σε σε περίπτωση καθυστέρησης ή άρνησης επιβίβασης ή ματέωση μιας πτήσης και δίνω αμέσω το λόγο στον κύριο Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε Κάλλα τη Επιτροπή, θα ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ την Κομισιόν για την πρωτοβουλία που έχει αναλάβει και την πρότασή τη για τα δικαιώματα των ε, επιβατών που πρέπει να προσαρμοστεί στην τωρινή κατάσταση. Όπω ξέρετε, δεν είναι ικανοποιητική η σημερινή κατάσταση σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά. Εδώ Πρόκειται για ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για τους πολίτες της Ευρώπης, ότι δεν τηρούνται τα δικαιώματα αυτά. Πολλές φορές η ευρωπαϊκή νομοθεσία για τους ε, Ευρωπαίους πολίτες φαίνεται να ξεπερνάει τα όρια αυτού που είναι απαραίτητο και άλλες φορές να περιορίζει τα δικαιώματά τους αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι θα υπάρξει μια σημαντική βελτίωση των δικαιωμάτων των πολιτών με τη θέσπιση περαιτέρω δικαιωμάτων που θα οδηγήσουν σε καλύτερη πληροφόρηση και άσκηση των δικαιωμάτων των ε, επιβατών των αεροπορικών εταιριών. Εγώ έχω λάβει υπόψη τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και τις σχετικές μελέτες είναι πάρα πολύ, ε, συνάντησα πάρα πολλούς εμπλεκόμενους επίσης από τον αεροπορικό κλάδο. Γι' αυτό που ήταν ιδιαίτερα σημαντικό για μένα είναι να υπάρχουν σαφείς και ε, κατανοήσιμοι κανονισμοί. Γι' αυτό έχω προσθέσει μερικές ακόμα πρόσθετες έννοιες στην πρόταση της Κομισιόν. Υπάρχουν ε, αεροπορικές εταιρείες οι οποίες δεν έχουν τηρήσει στο παρελθόν την, ε, τις υποχρεώσεις τους ή έχουν επικαλεστεί τεχνικά προβλήματα για κατάργηση ή καθυστέρηση ε, πτήσεων. Αυτά όμως δεν μπορούν να τύχουν επίκλησης όταν πρόκειται για εταιρείες που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Επιτροπή Μεταφορών κατάφερε να βελτιώσει σημαντικά την ε, πρόταση της Κομισιόν προς όφελος των επιβατών. Επίσης, σε ό,τι αφορά τα σημεία στα οποία τα κατόφλια από τα οποία ξεκινούν οι αποζημιώσεις, μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη υποστασία. Έχουν λοιπόν οι πολίτες δυνατότητα μετά από τρεις ώρες καθυστέρησης να έχουν, από... να έχουν 300 ευρώ αποζημίωση μέχρι αποστάσεως 3.500 600 ε, ε, ευρώ πάνω από, τις, <clears throat> πάνω από 3.500 χιλιόμετρα. Στο μέλλον θα πρέπει οι εταιρείε αεροπορικών εταιριών να δίδουν απάντηση σε όλα τα παράπονα των επιβατών και όχι να τα καθυστερούν για μήνε. Είναι λοιπόν απαραίτητη η βελτίωση των πληροφοριών και αυτό πρέπει να ξεκινήσει από τη διαδικασία κράτηση εισιτηρίων όπου υπάρχουν σαφή παράπονα και επίση η παροχή πληροφοριών στου αερολιμένε, όπου πρέπει να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο να μπορεί να δώσει σωστές πληροφορίες και να αντιμετωπίσει τα παράπονα των επιβατών. Είναι απαραίτητο επίσης να ενισχυθούν τα δικαιώματα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εγχείρημα για μας. Για την πολιτική no-show, μη παρουσία στο αεροδρόμιο, δεν θα πρέπει αυτό να δει δηλαδή σε άρνηση επιβίβαση στην πτήση επιστροφής, όταν δεν έχει πάει κανείς στην, πτήση, στην πρώτη πτήση. Επίσης και για την πτώχευση επιχειρήσεων έχουμε κάνει προτάσεις. Για τις πτήσεις τροφοδοσίας, η Κομισιόν έχει προτείνει η ευθύνη για την καθυστέρηση να, να ληφθεί υπόψη για την ευθύνη της εταιρείας η οποία τροφοδοτεί μια μεγαλύτερη πτήση η συνολική καθυστέρηση. Είναι απαραίτητο επίσης να έχουμε και πιο σαφείς κανόνες για τις χειραποσκευές και να απαγορευτεί η λογική ότι μόνο μία τσάντα θα μπορεί να επιβιβάζεται. Επίσης θα πρέπει να υπάρξουν οι απαραίτητες κυρώσεις στις αεροπορικές εταιρείες που δεν τηρούν τα, τους κανόνες και τα, για τα δικαιώματα των ε, ε επιβατών. Θέλω κατά τα άλλα να ευχαριστήσω τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων και τον εισηγητή της Επιτροπής ΙΜΚΟ και χαίρομαι για την ευκαιρία που έχουμε να συζητήσουμε τα θέματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Από την Κομισιόν έχει το λόγο ο κύριος Κάλλας. Κύριε Πρόεδρε, με αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κύριε Μπαχ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής Μεταφορών για το επικοδομητικό του έργο όσον αφορά την ρύθμιση αυτή. Στην πράξη, οι επιβάτες δεν καταφέρουν πάντα να επιβάλλουν τα δικαιώματά τους. Πρώτα απ' όλα γιατί το σύστημα επιβολής Τη Ρύθμιση που ισχύει σήμερα δεν είναι αρκετά αποτελεσματικό και δεύτερον γιατί δεν εφαρμόζεται το σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έπειτα, υπάρχει διαφορετική ερμηνεία του ίδιου κειμένου από πλευρά των επιβατών και από πλευρά των αερομεταφορέων. Η πρόταση τη Επιτροπή λοιπόν έχει ω στόχο να διευκρινίσει περισσότερο τα κείμενα και θέλει επίση να βελτιώσει και την επιβολή των δικαιωμάτων των επιβατών συγχρόνως ασχολείται με τις οικονομικές και λειτουργικές επιπτώσεις επί των αερομεταφορέων. Κάτι το οποίο σίγουρα βέβαια έχει επιπτώσεις και στην τιμή του εισιτηρίου για τους επιβάτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η πρόταση αυτή ενισχύεται από την Επιτροπή Μεταφορών σε διάφορους τομείς. Πρώτα απ' όλα στην επιβολή και δεύτερον στο δικαίωμα ενημέρωσης των επιβατών και επίσης και στο τι πρέπει να κάνει μια αεροπορική εταιρεία εφόσον ακυρωθεί μια πτήση και τι καταγγελίες προβλέπονται. Πάντως κάποιες από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μας προβληματίζουν. Ιδιαίτερα τα πρόκειται για τις καθυστερήσεις για τις μικρές και μεσαίες αποστάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να διατηρήσει τα τρέχοντα επίπεδα. Εσείς λέτε ότι μπορεί να είναι πολύ μικρά και ότι η ζημιά που έχουν οι επιβάτες είναι πραγματική. Δεν είναι εύκολο να βρούμε τον κανονικό χρόνο της καθυστέρησης, ποιος θα πρέπει να είναι αυτός, πάντως θα πρέπει να υπάρχουν κίνητρα για αποτροπή καθυστερήσεων. Εμείς θέλουμε οι επιβάτες να μπορούν να πάνε έγκαιρα εκεί που θέλουν να πάνε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει επίσης να εγκρίνει ένα εξελιτικό κατάλογο των έκτακτων περιστάσεων, των απρόβλεπτων καταστάσεων και να προβλέπονται ανάλογα οι αποζημιώσει. Εμεί πιστεύουμε ότι είναι πολύ περιοριστικό αυτό. Έπειτα το θέμα τη αφαιρεγκαιότητα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται τι ανησυχίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όμω, η πρόταση που λέει ότι οι αερομεταφορείς θα πρέπει να διαθέτουν είτε μια ασφάλιση είτε ένα ταμείο για να γίνεται επαναπατρισμό ή επιστροφή των χρημάτων των εισιτηρίων είναι ένα σύστημα το οποίο θα διπλασιάσει το κόστος. Δυσανάλογα μάλιστα. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 18 Φεβρουαρίου του 2013 όσον αφορά την περίπτωση αφιεγκαιρεότητας αναφέρει τις υποχρεώσεις που πρέπει να έχουν νερομεταφερεί και μπορούν να εφαρμοστούν πια. Ελπίζω κύριε Πρόεδρε ότι η σημερινή συζήτηση θα συνεισφέρει να βρούμε την σωστή ισορροπία ανάμεσα στα διάφορα συμφέροντα. Κύριος στόχος πάντως της Αναθεώρηση αυτής είναι καλύτερη επιβολή όσον αφορά τα δικαιώματα των ε, επιβατών, χωρίς βέβαια να πλήττονται τα κέρδη των αερομεταφορέων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Έχει το λόγο ο κύριος Χάνς Πέτρα Μάια. Έχετε το λόγο αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι πολύ σωστά τονίζει ο ισίτης ότι οι επιβάτες οι οποίοι για οποιοδήποτε λόγο χάνουν την πτήση ΑΛΕ, παραγωγός χάρη λόγω συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο, δεν πρέπει να χάνουν και την πτήση επιστροφής. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύσει όταν πρόκειται για μια πτήση με ανταπόκριση. Αν χάσει λοιπόν κάτι την πτήση ανταπόκρισης, χάνει τότε την πτήση επιστροφής. Αυτό θεωρώ ότι είναι λαθασμένο. Δεν πρέπει να εξαρτώνται τα δικαιώματα των επιβατών από το αν έχει κανείς μια πτήση με ανταπόκριση ή μια πτήση η οποία είναι κατευθείαν. Γιατί αυτό δημιουργεί μια ε, έλλειψη ίσης μεταχείρισης των ε, επιβατών. Κάποιο ο οποίο έχει πληρώσει ένα ειστήριο αλερετούρ λοιπόν δεν μπορεί να τύχει άρνηση να χρησιμοποιήσει την πτήση επιστροφή. Αυτό ήθελα να τονίσω από την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρο. Ακολουθεί ο κύριο Γκρό. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Α, κύριε εξαιρετικό κύριε πίτρο, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή τον ΣΟΣΠΑΚ γιατί νομίζω ότι έχει κάνει μια εξαιρετική εργασία η οποία έχει εξασφαλίσει ε, μια ισορροπία μεταξύ των αιτήσεων των επιβατών και από την άλλη μεριά των ε, συμφερόντων των αεροπορικών ε, εταιριών. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί πρώτα απ' όλα η διαφάνεια και αυτό ήταν το κύριο εγχείρημα το οποίο θέλουμε να έχουμε. Γιατί υπάρχουν οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που θα πρέπει να ενσωματωθούν πλήρως στην ε, νομοθετική ρύθμιση. Οι δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα είναι ότι υπάρχουν δυσκολίες με τη διαδικασία αποζημίωσης όταν παίρνει κανείς μια αποζημίωση 600 ευρώ για μια πτήση η οποία έχει ε, ακυρωθεί. Μπορεί αυτό να μην ικανοποιεί όμως τον επιβάτη γιατί έχει υποστεί μεγαλύτερη ζημιά. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έλαβε υπόψη του ο κύριος Μπαχ. Επίσης υπάρχει περίπτωση των ε, ε, φτηνών πτήσεων που κοστίζουν 20-30 ευρώ αλλά παίρνει μια αποζημίωση 600 ευρώ. Και αυτό το αντιμετωπίσαν στην Επιτροπή Μεταφορών. Επίσης το θέμα των έκτακτων συνθήκων. Νομίζω λοιπόν ότι όλα αυτά τα θέματα έχουν αντιμετωπιστεί και μπορεί να δώσει μια προστιθέμενη αξία αυτή η έκθεση όταν υπάρχει κοινό ορισμό του τι είναι οι έκτακτε συνθήκε και δεν υπάρχει διαμφισβήτηση. Το πιο σημαντικό για μένα όμω είναι η βελτίωση τη πληροφόρηση που δίνεται στου επιβάτε. Πριν κρατήσει κανεί μια θέση και η πληροφόρηση που μπορεί να έχει μετά στο αεροδρόμιο, ώστε να μην χρειάζεται κανείς να διαβάζει 20 σελίδες ψηλά γράμματα για να ξέρει πόσο μεγάλη μπορεί να είναι η βαλίτσα του. Επίσης, να υπάρχει και κάποιος, κάποια θηρίδα όπου μπορεί να υποβάλει παράπονα και να ζητήσει και να λάβει έγκυρες πληροφορίες. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία περιλαμβάνονται στην ε, έκθεση είναι θετικά για όλους και για μένα και για τις αεροπορικές εταιρείες και είναι μια επιτυχής ρύθμιση προς όφελος του Ευρωπαίου επιβάτη. Η κυρία Βερνιό έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα θα αποφασίσουμε για ένα σημαντικό κείμενο το οποίο θα προσφέρει πραγματική βελτίωση όσον αφορά τα δικαιώματα των συμπολιτών μας, οι οποίοι όλο και περισσότερο ταξιδεύουν με το αεροπλάνο και αντιμετωπίζουν συχνά δύσκολε καταστάσεις, είτε πρόκειται για την περιπλοκότητα των τιμών, είτε πρόκειται για την έλλειψη βοήθειας, είτε καταχρηστικών εμπορικών πρακτικών. Η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή περιλάμβανε έτσι κι αλλιώς πολλές βελτιώσεις σε σχέση με το σημερινό κείμενο. Νομίζω ότι καταφέραμε να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο και θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας και όλους τους συναδέρφους από τις άλλες ομάδες για το αποτέλεσμα αυτό αυτό. Προτείνουμε μια νομοθεσία που να μπορεί πραγματικά να εφαρμόζεται, γιατί δεν έχει νόημα να προσφέρουμε έκτενη δικαιώματα στους ε, επιβάτες, εάν μπορούν να ξεφεύγουν αεροπορικέ εταιρείε, είτε πρόκειται για τεχνικά ζητήματα, είτε για κανόνες οι οποίοι δεν είναι εφαρμόσιμοι. Γι' αυτό θέλουμε πολύ συγκεκριμένα να περιγράψουμε ποιε είναι οι απρόβλεπτες καταστάσεις. Επίσης, ο κανονισμός αυτός προσφέρει και μια σημαντική καινοτομία. Το δικαίωμα σε αποζημίωση αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρηση. Όμω πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι οι προορισμοί διαφέρουν μεταξύ του και άρα και οι ηλικοί περιορισμοί είναι διαφορετικοί και συγχρόνω πρέπει να έχουμε υπόψη μα ότι πρόκειται για έναν ενιαίο ευρωπαϊκό ενέργειο χώρο. Να έχουμε υπόψη μα επίση ότι πρόκειται για τρία διαφορετικά επίπεδα αποζημιώσεων. Εδώ πρέπει να στηρίξουμε βέβαια τι τροπολογίε οι οποίε είναι υπέρ των καταναλωτών, αλλά από την άλλη μεριά, το είπατε και εσεί κύριε Επίτροπε, κινδυνεύουν αεροπορικέ εταιρείε τελικά να ακυρώνουν μια πτήση αντί να προσπαθούν απλώ να έχουν μια καθυστέρηση. Επίση πρέπει να απαγορεύσουμε το να εμποδίζεται ο επιβάτη να μπει στο αεροπλάνο αν δεν έχει χρησιμοποιήσει το αλέ λόγω μιας ανταπόκρισης. Επίσης, οι τιμές πρέπει να είναι ξεκάθαρες για να μπορεί ο επιβάτης να συγκρίνει την κατάσταση, όπως και το δικαίωμα για να μεταφέρει αποσκευές τόσο στην καμπίνα όσο και στον ειδικό χώρο αποσκευών. Και πρέπει οι αεροπορικές εταιρείες να προβλέπουν σήμερα επαφή στα διάφορα αεροδρόμια αν υπάρξει πρόβλημα. Έχουμε ένα ισορροπημένο κείμενο ανάμεσα στα δικαιώματα που είναι ισορροπημένα για του επιβάτε και από την άλλη μεριά τι υποχρεώσει που είναι ρεαλιστικέ για τι επιχειρήσει. Ελπίζω να έχουμε μια καλή συζήτηση με το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. κυρία Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριε Κάλλας, συναδελφοί για την ομάδα των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων και Δημοκρατών ήθελα να πω ότι εμείς πάντα υποστηρίζαμε τα δικαιώματα των επιβατών. Εγώ έχω συνεργαστεί σε πολλές εκθέσεις που αφορούσαν το θέμα αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαιώματα αυτά. Η σημερινή έκθεση προέκυψε λόγω των συχνών περιστατικών ακύρωσης πτήσεων, μεγάλων καθυστερήσεων ή παρατυπιών στο χειρισμό των αποσκευών. Μόνο το 2% των επιβατών λαμβάνουν την αποζημίωση την οποία δικαιούνται το νέφος που προέκυψε με τη, από το υφέστο της Ισλανδίας ε, κατέδειξε την ανάγκη να υπάρξει ένα καλύτερο πλαίσιο για τα δικαιώματα των επιβατών και τις υποχρεώσεις των αερομεταφορέων οι επιβάτες πρέπει να ενημερώνονται σωστά και πρέπει να υπάρχει ένα σωστό σύστημα αποζημίωσης. Είναι πολύ σημαντικό οι επιβάτες να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Σήμερα, πολύ συχνά, οι επιβάτες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Και οι αερομεταφορείς ε, δεν τους ενημερώνουν επαρκώς. Καλωσορίζω το γεγονό ότι τώρα, χάρη στη δουλειά τη Επιτροπή Μεταφορών, έχουν το δικαίωμα αποζημίωση ή επιβάτε σε περίπτωση ακύρωση ή καθυστέρηση. Όσον αφορά του ανθρώπου με προβλήματα κινητικότητα, στο μέλλον θα υπάρχει εκπαίδευση των πληρωμάτων, θα υπάρχουν σκυλιά καθοδήγηση και δεν θα είναι πλέον δυνατόν να αφαιθούν ε, πίσω άνθρωποι με αναπηρία απλά και μόνο διότι δεν συνοδεύονται. Καλωσορίζω το γεγονό ότι η Επιτροπή Μεταφόρων υποστήριξε τις περιφερειακές αεροπορικές εταιρείε και το χρόνο αυτό των 90 λεπτών κατά τον οποίο δεν θα έχουν υποχρέωση αποζημίωσης για ε, απώλεια της, ε, ε, της ανταπόκρισης. Καλωσορίζω και το γεγονό ότι οι επιβάτε θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πτήση επιστροφή ε, όταν ε, δεν έχουν χρησιμοποιήσει την πτήση Αλλά Λυπούμε για τη συμπεριφορά τη ομάδα των Σοσιαλιστών, η οποία υποστήριξε όλε τι συμβιβαστικέ στην Επιτροπή. Αλλά τώρα προσπαθεί να τι άρει. Γι' αυτό το λόγο εμείς ε, στο ΑΛΔ δεν υποστηρίζουμε τις τροπολογίες Μάιερ Τελικά θα ήθελα να αναφέρω και το πρόβλημα του Γιβραλτάρ. Παρακαλώ περατώστε αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ τον εισήγητη για την εξαιρετική συνεργασία. Είναι μεγάλο ο κατάλογο των αγορητών και έχουμε στη συνέχεια ψηφοφορίε. Γι' αυτό παρακαλώ όλου του συναδέλφου να παραμείνουν μέσα στα όρια του χρόνου αγόρευση. Ο κύριο Τέιλα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Έρχομαι να σας μιλήσω σήμερα ως εισηγητής στην περσινή έκθεση για τον κανονισμό 261 του 2008 και ως κοιόδης των Πρασίνων για την έκθεση του κυρίου Μπαχ σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο εισηγητή για την επικοδομητική του προσέγγιση. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να πω ότι καταφέραμε να αλλάξουμε το επίκεντρο στην πρόταση της Κομισιόν από μια τάση υποστηρίξης της βιομηχανίας, του τομέα και των αερομεταφορέων σε μια προσέγγιση που υποστηρίζει περισσότερο τους επιβάτες. Παρότι η άποψη της ομάδας μου ήταν ότι η αποζημίωση πρέπει να καταβάλλεται μετά από μια ώρα, δεν έγινε δεκτή. Το όριο των τριών ωρών έγινε δεκτό και αυτό αντικατοπτρίζει και την αποφάση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το, ότι τρεις ώρες θα είναι το σημείο ενεργοποίησης. Είναι πολύ καλύτερη λοιπόν η κατάσταση σε σχέση με την αρχική θέση της Κομισιόν που ήταν ε, πέντε ώρες. Επίσης καταφέραμε να υποστηρίξουμε το περιορισμό των εξαιρετικών περιστατικών ώστε να σταματήσουν οι αερομεταφορείς ε, να χρησιμοποιούν αυτή την αιτιολογία ώστε να αποφεύγουν να καταβάλουν αποζημιώσεις σε επιβάτες που τις δικαιούνται. Χαίρομαι που βλέπω τη σύσταση για καλύτερη ενημέρωση των επιβατών και ελπίζω ότι η υλοποίηση θα μπορέσει να βελτιωθεί. Για αυτό το σκοπό η πρότασή μας ανεξάρτητων οργανισμών μεσολάβησης ε, πιστεύω θα αποδειχθεί εξαιρετικά ωφέλιμη. Επίσης η διάταξη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την ενεργειακή απόδοση των ταξιδιών των επιβατών θα, βρίσκονται, θα αναγράφονται στους ιστότοπους και στα εισιτήρια των ταξιδιωτών. Δεν μπορούμε να αναμένουμε από τους ανθρώπους να δείχνουν ευθύνη όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα όταν δεν γνωρίζουν ποιες είναι οι επιπτώσεις. Χαίρομαι που μπόρεσα να υποστηρίξω αυτήν την εκτίση και θέλω να την ευχαριστήσω τον κύριο Μπάχ για την επικοδομητική του προσέγγιση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank Ευχαριστούμε κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ήδη από το 2004 με την ομοθεσία εκεί με εισηγητή από το ΕΛΚΑ προσέφερε αρκετά πλεονεκτήματα για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών. Όπως σωστά αναφέρθηκε μετά από την ιστορία με τον νέφος του Ισλανδικού ηφαιστείου, Καλά κάνουμε που ξανακοιτάμε την νομοθεσία ώστε να επιφέρουμε μια καλύτερη ισορροπία. Ευχαριστώ λοιπόν τον εισηγητή, τον κύριο Πάχ, ο οποίος προσπάθησε να βρει μια καλή λύση. Και σίγουρα μετά από αυτή τη δουλειά που έριξε αξίζει καλές διακοπές. Άλλαξαν κάποια πράγματα σε σχέση με την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα έχουν επιπτώσεις επί των επιβατών. Εγώ πιστεύω ότι κινδυνεύουμε να αυξήσουμε έτσι τις τιμές και να περιορίσουμε την επιλογή των επιβατών. Υπάρχουν βέβαια πλέον εκτήματα και το ότι άλεξε το θέμα των 90 ε, λεπτών, ότι είναι πιο σαφές το θέμα της ενημέρωσης και ότι πιο εύκολα μπορούν να κάνουν καταγγελίες και να έχουν αποζημιώσεις οι επιβάτες. Έπειτα υπάρχουν όμως τα περιφερειακά αεροδρόμια, τα οποία δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Όμως αν εγκριθεί η έκθεση αυτή, κινδυνεύει εκεί να δημιουργηθεί πρόβλημα για αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια. Το ότι άλλαξε το 5 και έγινε 3 ώρες. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερες ακυρώσεις και αυτό θα ήταν λυπηρό. Άρα τελικά τα feeder flights μπορεί να περιοριστούν και να καταστραφούν διάφορες συμφωνίες ε, για μεγάλες πτήσεις με που κάναμε δεκαετίες να τα φτιάξουμε. Τα επίπεδα αποζημίωσης τώρα δεν αντικατοπτρίζουν συχνά το κόστος των φτηνών εισιτηρίων που πολλές φορές έχει ο κόσμος. Εγώ θα ήθελα εκεί το κόστος να εξαρτάται, δηλαδή το κόστος αποζημίωσης, από το τι πληρώνει κανείς για το εισιτήριό του. Πολλά από αυτά τα θέματα ελπίζω να μπορέσουν να λυθούν. Τέλος, έχω υποβάλει διάφορες τροπολογίες όσον αφορά το Γιβραλτάρ. Στην αρχική ρύθμιση υπήρχαν, ζήτησαν να αφαιρεθούν, δεν έγινε όμως. Το 2006 οι κυβερνήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου της Ισπανίας και Γιβραλτάρ υπέγραψαν συμφωνία που σημαίνει ότι το Γιβραλτάρ αποτελεί μέρος της ενιαίας αγοράς είναι Βρετανική επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να επεκταθούν και εκεί τα ίδια δικαιώματα όπως οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ισχύουν. Χάσαμε στην Επιτροπή Μεταφορών την ψηφοφορία, αλλά έχω υποβάλει εκ νέου τις τροπολογίες αυτές και ελπίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να με στηρίξει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κόλιτσεκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, τα δικαιώματα των επιβατών ρυθμίζονται εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μόνο τα τελευταία χρόνια προωθούνται περισσότερο στα αεροδρόμια. Με τη σχετική ενημέρωση, οι επιβάτες έχουν τρεις μήνες για να υποβάλουν καταγγελίες ε, σε αερομεταφορέα. Εντός δύο μηνών πρέπει να έχει λαβεί ο επιβάτης απάντηση μετά από μια καταγγελία. Αυτό που έχουμε εδώ είναι μια, ένα συμβιβασμό ε, που προσπαθεί να αποτρέψει τους αερομεταφορείς να αποφεύγουν τις ευθύνες τους ε, προς το επιβατικό κοινό. Υπάρχει ένας ε, μη εξαντλητικός κατάλογος εξαιρετικών περιστάσεων. Το παράρτημα 2 είναι ένα απλό εγχειρίδιο για τους επιβάτες Διάφορα ζητήματα έχουν βελτιωθεί σε σχέση με το 2004 όσον αφορά τα μικρά παιδιά, τους ανθρώπους με αναπηρίες ή τους επιβάτες που μεταφέρουν μουσικά όργανα. Στο μέλλον, σε περίπτωση εισιτηρίων με πολλαπλές ανταποκρίσεις, ε, οι επιβάτες θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένες, αλλά όχι όλες τις πτήσεις που έχουν κρατήσει. Επίσης ε, καταφέραμε έναν ισορροπημένο συμβιβασμό όσον αφορά την τιμολόγηση. Αυτό είναι ένα νέο πρότυπο για την ε, αεροπλοεία. Θα επιθυμούσα να ε, πω στον κύριο Επίτροπο ότι στην Τσεχική Δημοκρατία τα ταξιδιωτικά πρακτορία έχουν είναι ασφαλισμένα κατά της αφαιρεγγιότητας. Πάλι ξεπερνάτε το χρόνο ομιλή σας, παρακαλώ ή να μην το πράτετε, η κυρία Ντότη έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ παρούσα η κυρία Ντότ, ο κύριος Κόχ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έκθεση του συναδέλφου μου του κυρίου Γκέορκ Μπαχ έχει επιτύχει μια σωστή ισορροπία μεταξύ των συμφερόντων των αεροπορικών εταιριών και των δικαιωμάτων των επιβατών. Αν λάβουμε υπόψη τη σημερινή κατάσταση και επίσης την πρόταση της Κομισιόν υπάρχει μια σημαντική βελτίωση. Υπάρχει ένας κίνδυνος ότι αν θέλετε να ε, βοηθήσετε τους ε, επιβάτες θα πρέπει να σταθούμε κάπως κριτικά σε σχέση με τις τροπολογίες. Είναι ορισμένες τροπολογίες τις οποίες εγώ ζητώ να απορριφθούν παραδείγματο χάρη αυτές που θεσπίζουν την ε, έννοια των κατοφλίων για την ε, ε, αποζημίωση. Εμείς με δύο κατόφλια έχουμε δώσει τη δυνατότητα στις εταιρείε να ε, έχουμε δώσει δύο κατόφλια για τις εταιρείε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος οι αεροπορικές εταιρείε να καταργούν πτήσεις αντί να πληρώνουν την αποζημίωση. Επίσης φοβόμαστε ότι οι αεροπορικές εταιρείε ότι θα λάβουν υπόψη τον κίνδυνο να πληρώσουν αποζημιώσεις λόγω της νέας νομοθεσίας και θα ενσωματώσουν το κόστος, θα το μετακυλήσουν στον καταναλωτή. Είναι απαραίτητο λοιπόν να δώσουμε στις αεροπορικές εταιρείες να έχουν καλύτερες προτάσεις προς τους επιβάτες. Οι επιβάτες θα κερδίσουν από κάτι τέτοιο. Αν δεν μπορεί όμως μια αεροπορική εταιρεία λόγω αυτής της νομοθεσίας να δίνει ε, ευνοϊκές προτάσεις και προσφορές, τότε θα βγει από την αγορά. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τη μακροχρόνια υγεία των αεροπορικών εταιριών και όχι μοναχά το βραχυπρόθεσμο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει μια μπλε κάρτα προς εμάς. Ο κύριος Λάιτφριτ θέλει να σας θέσει ένα ερώτημα. Το δέχεστε κύριε Κόχ. Κύριε Λάιτφριντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κόχ. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον αυτά που είπατε. Ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μεγαλύτερη ε, προσοχή προς τις ανάγκες των εταιριών και όχι των καταναλωτών. Αυτή είναι η θέση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Θέτουμε τους πολίτες και τους καταναλωτές σε δεύτερη μοίρα. Σας κατάλαβα καλά ή όχι, κύριε Κόχ η πολιτική είναι μια εξισορρόψη συμφερόντων. Με καταλάβατε σωστά. Πρέπει να ληφθούν υπόψη και τα συμφέροντα και το δύο πλευρό, λέει ο κύριο Κόχ. Ακολουθεί ο κύριο Ελ Χαδραουί. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αγαπητοί συνάδελφοι. Σήμερα εξετάζουμε μια σημαντική υπόθεση που βοηθάει τους καταναλωτές με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και διευκρινίζει τα δικαιώματά τους. Ο οργανισμός του 2004 χρειαζόταν αναθεώρηση. Ακριβώς γιατί άφηνε πολλά παραθυράκια ανοιχτά για καταχρήσεις. Και δεν υπήρχε πάντα απόδοση δικαιοσύνης. Τώρα με τον εισηγητή Μπαχ και με την ε, βοήθεια των σκιωδών εισηγητών και των υπολείπων συναδέρφων έχουμε ένα κανονισμό πολύ πιο συγκεκριμένο. Το δικαίωμα στην αποζημίωση πια υπάρχει και σε περίπτωση καθυστερήσεων, όχι μόνο ακύρωσης και διευκρινίστε πολύ καλύτερα το ποιε είναι οι απρόβλεπτες καταστάσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό να περιλαμβάνεται στην νομοθεσία. Σημαντικό επίσης είναι ότι προβλέπεται και βοήθεια προς τους επιβάτες εφόσον υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο αεροδρόμιο και υπάρχει και υποχρέωση της ενημέρωσης αν κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, προβλέπεται το τι ε, δικαιώματα έχουν οι επιβάτες, πώς γίνονται οι καταγγελίες, τι αποσκευές μπορούν, έχουν δικαίωμα να μεταφέρουν στο αεροσκάφο, στην καμπίνα κλπ. Αν συγκρίνουμε δηλαδή τώρα την πρόταση της Επιτροπής με τον κανονισμό που υπάρχει, και τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι πια έχουμε σαν κάτι πολύ ενδιαφέρον πάνω στο οποίο να δουλέψουμε. Αποτελεί πρόοδο και βοηθούνται οι επιβάτες τους οποίους θέλουμε πάντα να εξυπηρετούμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Ντότ είναι παρούσα τώρα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε εκτιμώ ιδιαίτερα που μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ως βουλευτής που εκπροσωπώ τη Βόρεια Ιρλανδία που βρίσκεται στην περιφέρεια της Ευρώπης γνωρίζω τα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι πολίτες της χώρας μου λόγω των μακρών καθυστερήσεων και καμιά φορά των ακυρώσεων πτήσεων. Χαιρετίζω λοιπόν αυτή τη συζήτηση για την καλύτερη προστασία των πολιτών. Για να μπορούμε να έχουμε οικονομική ανάπτυξη πρέπει να ενθαρρύνουμε το επιχειρήν και τις επιχειρήσεις και την αύξηση του τουρισμού. Ένα σημαντικό τμήμα αυτού του εγχειρήματο είναι να το εξασφαλίσουμε ότι η εργατική μας δύναμη και οι επισκέπτες νιώθουν εμπιστοσύνη όταν ταξιδεύουν με αεροπορικές ε, εταιρείες. Η το νομοθέτημα αυτό θα εξασφαλίσει ότι οι επιβάτες οι οποίοι υφίστανται μακρές καθυστερήσεις θα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα θύματα ακυρώσεων. Και επίσης επεκτείνει το δικαίωμα για την παροχή στέγαση σε αυτές τις περιπτώσεις και δίνει και δικαιώματα στους επιβάτες που έχουν μειωμένη κινητικότητα. Επίσης υπάρχει καλύτερη προστασία σε περίπτωση πτώχευση αεροπορικών εταιριών. Όλα αυτά είναι θετικά. Πρέπει να αναγνωρίσουμε όμως ποιε είναι και οι ευκαιρίες που θα πρέπει να δημιουργηθούν για το όφελος των περιφερειακών οικονομιών και των αεροπορικών εταιριών του για τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι όταν προστατεύουμε του επιβάτε δεν θέτουμε υπερβολικό άχθο στι επιχειρήσει με την νομοθεσία και τη ρύθμιση. Γιατί πρέπει αυτέ οι εταιρείε να μπορούν να κάνουν επενδύσει και να προοδεύσουν. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μάση να έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, αγαπητέ Τζόρτζ, και εσύ κάνει μια εξαιρετική εργασία και είναι πραγματικά ένα πολύ μεγάλο βήμα για τους επιβάτες αεροπορικών εταιριών σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων. Όλοι ξέρουμε τι μπορεί να γίνει. Μπορεί να χάσει κανεί βαλίτσε, μπορεί να έρθει το αεροπλάνο να ανταπόκριση πολύ αργά. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να πάνε στραβά και τα έχουμε ζήσει όλα. Γι' αυτό είναι αποφασιστικό να υπάρξει μια βελτίωση. πρόταση έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα από την έκθεση του George Bach που είναι ακόμα πιο φιλική για τους ε, επιβάτες και γι' αυτό πρέπει να την υποστηρίξουμε. πέτυχε σημαντικές βελτιώσεις. Καλύτερη, ε, σοβαρότερη αποζημίωση σε περίπτωση καθυστέρησης και επίσης να μπορεί κανείς να αποζημιώνεται στον τόπο άφηξης και όχι μόνο στον τόπο εκκίνησης έχουμε εξασφαλίσει να υπάρχει καλύτερη πληροφόρηση για όλους τους επιβάτες, το οποίο εξασφαλίζει και τη διαφάνεια και το γεγονός ότι θα υπάρχει πάντα κάποιος συνομιλητής του επιβάτη, ο οποίος μπορεί να δεχτεί παράπονα και να δώσει πληροφορίες. Πολλές φορές αυτό δεν συμβαίνει. Έχουμε τη δυνατότητα επίσης να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια ό,τι αφορά τη μεταφορά μουσικών οργάνων και επίσης και το θέμα των αποσκευών. Ο κανόνας αυτός ότι μόνο ε, μια βαλίτσα μπορεί να έχει κανείς. Αυτό πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα για επιβάτες οι οποίοι έχουν να κάνουν υπερατλαντικές πτήσεις και δεν μπορούν να περιοριστούν σε μια, σε μια βαλίτσα. Επίσης, πιστεύω πρέπει να εξασφαλίσουμε όλα αυτά τα δικαιώματα. Έχετε μια μπλε κάρτα κυρία... Κυρία Λίχτεμπεργκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. έχω χρησιμοποιήσει το χρόνο μέχρι την απόφαση που επίκειται για να δω τι γίνεται στις ε, πτήσεις ανταπόκρισης και να ρωτήσω επιβάτες αν έχουν πάρει αποζημίωση σε περιπτώσεις καθυστέρησης, αν την έχουν ζητήσει ή αν την έχουν πάρει πράγματι. Είναι απογοητευτικά τα αποτελέσματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν κάνουν καμία διεκδίκηση γιατί θεωρούν ότι δεν πρόκειται να πάρουν τίποτα, αλλά και αυτοί οι οποίοι έχουν διεκδικήσει κάποια ε, αποζημίωση με πολύ δυσκολία μπορούν να αποκομίσουν κάποια πραγματική αποζημίωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ υπενθυμίζω ότι ο κύριος Κάλλας έχει υποβάλει μια πρόταση η οποία φαίνεται να έχει κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει από ό,τι φαίνεται μονάχα α, αντιμετωπίσει τις ανάγκες των αεροπορικών επιχειρήσεων και όχι των επιβατών. Αυτό το οποίο με ενοχλεί ακόμα περισσότερο είναι η έννοια της ανωτέρα βία έχει διατυπωθεί με τέτοιο τρόπο ώστε μπορεί χάρη στην περίπτωση τέφρας από ηφαίστειο που έλαβε χώρα πριν από δύο χρόνια να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ενός επιβάτη να ζητήσει αποζημίωση για το παραμικρό. Η Επιτροπή Μεταφορών και η Επιτροπή Εσωτερικής Αγορά έχουν εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα των επιβατών έχουν βελτιωθεί. Γι' αυτό ζητώ την υποστήριξή σα για τι τροπολογίε που έχουμε καταθέσει. Τονίζω ότι είναι σαφέ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τα δικαιώματα των επιβατών γιατί βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μονοπωλιακή δομή η οποία δεν δίνει πεντάρα για του επιβάτε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λίχτεμπεργκ. Έχετε μια μπλε κάρτα, τον κύριο Κράμερ. Χωρίς μικρόφωνο κύριος Κράμερ. για τον κανόνα της μίας βαλίτσας. Μήπως είναι μία διάκριση εναντίον των, των χειραποσκευών, συγγνώμη, για εναντίον των γυναικών. Όταν είμαι μία γυναίκα και έχω και μία μικρή τσάντα μαζί μου, πρέπει να πληρώσω. Ενώ ένας άντρας δεν μπορεί δεν, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Μήπω είναι μια διάκριση λοιπόν κατά των γυναικών αυτό, το γεγονό ότι οι άντρε δεν κουβαλάνε τι αντούλε αυτού του είδου, κυρία Λίχτεμπεργκερ. Είναι μια διάκριση για όλου αυτού είτε είναι άνδρες είτε είναι γυναίκες, αλλά φυσικά αφορά πολύ περισσότερο τις γυναίκες οι οποίες πρέπει να αλλάξουν, όταν πρέπει να αλλάξουν πτήση και πολλές φορές θα πρέπει να πάρουν την, ε, την τσάντα τους μαζί για να μην χάσουν την επόμενη πτήση. Έχω χάσει τη βαλίτσα μου πάρα πολλές φορές σε ανταποκρίσεις και αυτό μου δημιουργεί δυσκολίες. Γι' αυτό πάρα πολλοί προσπαθούν να έχουν μαζί τους τις ε, αποσκευές τους για να είναι σίγουροι ότι θα μπορέσουν να την έχουν τη βαλίτσα τους και στον προορισμό τους. Ο κύριος Μπράντμπερν έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τους τελευταίους μήνες στο κοινοβούλιο αυτό είχαμε την ευκαιρία να προβούμε σε μια μακροχρόνια βιώσιμη βελτίωση στις ζωές ε, των ε, πολιτών μας. Κάποιες αεροπορικές εταιρείες αποκρύπτουν τα δικαιώματα από τους επιβάτες για αρμόζουσα αποζημίωση σε περίπτωση σημαντικών καθυστερήσεων στα ταξίδια τους. Με την αναθεώρηση αυτού του κανονισμού και τη νέα ολοκληρωμένη λίστα των εξαιρετικών περιστάσεων κλείνουμε τα παραθυράκια τα οποία δεν επέτρεπαν στους επιβάτες ε, να λάβουν αποζημίωση σε περίπτωση καθυστερήσεων των αερομεταφορέων λόγω κακής ε, διαχείρισης. Στο μέλλον οι επιβάτες θα λαμβάνουν καθαρές πληροφορίες όσον αφορά τα επιτρεπόμενα βάρη αποσκευών και θα είναι βέβαιο πλέον ότι δεν θα παρεμποδίζεται να ψωνίζουν σε αεροδρόμια από του αερομεταφορεί. Παρά όλα αυτά τα δικαιώματα των επιβατών, ε, υπάρχει μια εξαίρεση. Το Γιβραλτάρ, αν οι τροπολογίε ε, που αναγνωρίζουν το Γιβραλτάρ ε, ω ευρωπαϊκό αεροδρόμιο δεν περάσουν, δεν θα μπορέσω να υποστηρίξω αυτή την νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ομάζη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, δεν θα μακρηγορήσω, ήθελα απλά να επιστήσω την προσοχή εδώ της συνέλευσης ε, στην μεταχείριση προς τους επιβάτες που έχουν ως προορισμό ή που προέρχονται από τις άκρως απόμακρες περιοχές. Αυτές οι πτήσεις στον κανονισμό θεωρούνται εξοκοινωτικές κατά όλων των αρχών ε, σύμφωνα με τις οποίες οι άκρως μακρές περιοχές ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απορρέει από αυτό φυσικά ε, ένα λίγο ευνοϊκό καθεστώς αποζημιώσεων σε περίπτωση καθυστερήσεων. Πρέπει λοιπόν να υποβάλω κάποια σειρά τροπολογιών για να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση και καλό τους συναδέλφους να τις υποστηρίξουν. Ευχαριστούμε. Ο ε, κύριος Ντάρτμουθ. Έχω την τιμή να εκπρόσωπω το Γιβραλτάρ και το λαό του. Και αυτή τη στιγμή ομιλώ για να αντιμετωπίσουμε τα πιθανά προβλήματα στο αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ. Η κατάσταση έχει ως εξής. Η κυβέρνηση της Ισπανίας ε, συστηματικά και όπως βλέπω εγώ εκδικητικά επιβάλλει μικροελέγχους ε, στα χερσαία σύνορα μεταξύ Γιβραλτάρ και Ισπανίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μαζικές ε, απαράδεκτες καθυστερήσεις. Και μάλιστα αυτοί που υποφέρουν από αυτέ τι καθυστερήσει είναι περισσότερο Ισπανοί πολίτε. Λόγω των προβλημάτων στα χερσαία σύνορα, η, τα αεροπορικά ταξίδια γίν, αποκτούν ύψιστη σημασία. Και οι προσπάθειες που γίνονται από μέλη του Κοινοβουλίου αυτό μέσω νομοθεσιών να καταπνίξουν τις αερομεταφορές προς και από το αεροδρόμιο του Γιβραλτάρ δεν μπορούν να συνεχιστούν. Είναι κάτι απαράδεκτο και σας παρακαλώ να υποστηρίξετε τις τροπολογίες μου σήμερα να τονίσω ότι Thank you. Do you accept the blue card? Α, δέχεστε μια μπλε κάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βουλευτά, δεν θυμόσαστε καλά τα πράγματα για το Γιβραλτάρ, διότι το τα συμβάντα πας που γίνονται στα σύνορα, στο πέρασμα δηλαδή, ανάμεσα στην ε, γραμμή του Γιβραλτάρ, είχε να κάνει με επιθεωρητές ε, της Κομισιόν, οι οποίοι βλέπαν τι γίνεται με την εφαρμογή του Σέγγεν. Εσείς ξεχνάτε τα συμπεράσματα των επιθεωρητών που είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, υπάρχει ισορροπία και υπάρχει μια υποχρέωση ελέγχου για να μην υπάρχει λαθρεμπόριο. Ευχαριστούμε κύριε Γκράντε Στεπάσκο. Ο συνάδελφος Ντόρμουτ. Να σας διαβεβαιώσω ότι η μνήμη μου είναι πάρα πολύ καλά. Και μάλλον καλύτερα από τη δικιά σας. Ναι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήγε και επιθεώρησε. και ανοήτως ενημέρωσε την Ισπανική κυβέρνηση έξι εβδομάδες πριν. Οπότε οι Ισπανικές αρχές, για να το πω ευγενικά, διόρθωσαν την κατάσταση για την επίσκεψη αυτή. Εσείς και οι συνάδελφοί σας θα έπρεπε να ντρέπεστε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Δικέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να Ευχαριστώ τον συνάδελφο Μπαχ για την πρόταση αυτή. Η πρόταση αυτή λοιπόν εξετάζει τα δικαιώματα των ε, επιβατών σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση, ακύρωση, πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση και μάλιστα οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου ενισχύουν τα δικαιώματα των ε, επιβατών ε, μέσω των τροπολογιών του ίδιου του συγκεκριτή αλλά και των ευρωβουλευτών. Έτσι λάβαμε υπόψη μας την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πλέον ο νομοθέτης έπρεπε να ασχοληθεί και να μην προστίθεται στο άγχος που έχει ο επιβάτης από το ταξίδι ένα επιπλέον άγχος στην περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Αναφέρουμε λοιπόν ποιες είναι οι περιπτώσεις και πολύ συγκεκριμένα όπου έχει δικαιώματα αποζημίωσης ο επιβάτης. Τώρα με τις τροπολογίες μας ενισχύονται λοιπόν τα δικαιώματα αυτά και προβλέπονται και ειδικά έντυπα για καταγγελίες και συγκεκριμένος τρόπος εφαρμογής των κειμένων. Όμως με στεναχωρεί το εξή, ότι δεν καταφέραμε να πείσουμε τους συναδέρφους να περάσουν την ε, διάταξη που απαγορεύει σε μια αεροπορική εταιρεία να μην επιτρέψει την επιβίβαση ενός επιβάτη επειδή έχει χάσει το αλέ και δεν το επιτρέπει να πάει ε, στη συνέχεια της πτήσης. Δεν θα έπρεπε το δικαίωμα αυτό να το χάνει ο επιβάτης για εμπορικούς λόγους. Η απαγόρευση επιβίβασης πρέπει να έχει να κάνει μόνο με περιπτώσεις ασφάλειας ή έκτακτες συνθήκες, είτε υγειονομικού χαρακτήρα ή για λόγους τρομοκρατίας. Αν αρνείται την επιβίβαση μια αεροπορική εταιρεία αυθαίρετα, τότε θα πρέπει να μπορεί να το καταγγείλει αυτό ο επιβάτης και να κερδίζει. Ελπίζω να μην υπάρξουν συνάδελφοι οι οποίοι θα βρεθούν σε αυτή την κατάσταση και τότε να μετανιώσουν που δεν πέρασαν την πρόβλεψη αυτή. Ζητώ την κατανόησή σας για το γεγονός ότι δεν μπορώ να λάβω κανένα, καμία αίτηση για μπλε κάρτα γιατί έχουμε περάσει και έχουμε καθυστερήσει με το χρόνο των ομιλητών. Δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Δεν έχουμε λοιπόν τη δυνατότητα να ακούσουμε περαιτέρω ερωτήσεις με μπλε κάρτα. Ακολουθεί η κυρία Γιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δέκα χρόνια είμαστε σήμερα μετά τον πρώτο κανονισμό για τα δικαιώματα των επιβατών. Μιλάμε λοιπόν για την αναθεώρηση. Έχουμε κάνει κανονισμού για τους επιβάτες σιδηροδρόμων κλπ. Χαίρομαι λοιπόν που επιπλέον ασχολούμαστε με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για την ευκολία με την οποία πρέπει να προβαίνουν σε καταγγελίε οι επιβάτε και χάρη στον εισηγητή Μπαχ που έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία καταφέραμε να ασχοληθούμε και με τα άτομα με ειδικέ ανάγκε οι οικογένειε με μικρά παιδιά που έχουν τα καροτσάκια και να μπορούν να πηγαίνουν πηγαίνουν μέχρι την πόρτα του αεροπλάνου με αυτά ή τα άτομα που έχουν αναπηρική καρέκλα και αυτοί να μπορούν εύκολα να μπαίνουν στο αεροπλάνα. Ή μιλάμε επίσης και για τους επιβάτες μουσικούς που έχουν μουσικά όργανα μαζί τους και να μπορούν πλέον να τα έχουν στην καμπίνα. Υπάρχουν πολλές ε, τροπολογίες λοιπόν θετικές υπέρ των ατόμων αυτών είτε με αναπηρία είτε οικογένειες με μικρά παιδιά που όπως είπα μπορούν με τα καροτσάκια να φτάσουν μέχρι την είσοδο του αεροπλάνου. Υπάρχει και η ρύθμιση που λέει ότι δεν μπορεί κανείς να έχει την τσάντα όπω οι κυρίες που κυκλοφορούν με την ε, τσάντα. Εκτός από την χειραποσκευή που έχουν δικαίωμα να φέρουν μέσα στην καμπίνα του αεροπλάνου, μπορούν να έχουν και αυτή την τσάντα. Χαιρόμαστε λοιπόν που υπάρξει ενημέρωση του κανονισμού αυτού που είναι και αποτρεπτική για αεροπορικές εταιρείες που θέλουν να κάνουν καταχρήσεις. Μιλάμε επίσης για την αφαραγκαιότητα, μιλάμε για την πάυση δραστηριοτήτων αεροπορικών εταιριών που αφήνουν καθυλωμένους τους επιβάτες ε, στο εξωτερικό. Και υπάρχουν και άλλες τροπολογίες που μιλάνε για τις αποζημιώσεις προκειμένου αυτές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές καταστάσεις, δηλαδή να αλλάζουν τα ποσά κάθε τόσο. Οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει επίσης να εξυπηρετούν τους πολίτες, να τους στείλουν νερό για παράδειγμα, να πάσα στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Μάισνερ, έχετε δίκιο. Δεν, δεν Είδα ότι θέλατε να θέσετε ένα ερώτημα. Έχετε το λόγο λοιπόν. Χωρίς μικρόφωνο. Ήθελα να θέσω ένα ερώτημα στον κύριο Ρικέ προηγουμένως. Ντομινίκ. Ε, Ντομινίκ, θέλω να σου θέσω ένα ερώτημα. Μια μπλε κάρτα. Κύριε Ρικέ, δέχεστε την ερώτηση της κυρίας Μάισνα. Κύριε Ρικέ, λοιπόν. Αναφέρθηκε το θέμα της ε, εχθρότητος προς τις γυναίκες σε σχέση με τον κανόνα με τη μία χείρα Εμείς θεωρούμε ότι μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα με αυτή την νομοθετική πρόταση, να υπάρξει άρση της διάκρισης. Αυτό ήταν ακριβώς το, ο στόχος μας. Και πιστεύω ότι το έχετε κατανοήσει ότι αυτό θέλαμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ κύριε Ρικέ. Φυσικά συμμερίζομαι την παρατήρηση του θέματος Φυσικά πρέπει να δούμε τι εννοούν ε, οι συναδελφοί γυναίκες με την τσάντα χειρός ε, ε, γιατί πολλές φορές μπορεί να μοιάζει με βαλίτσα. Συνεπώς υπάρχει περιθώριο διαφόρων αρμενιών. Αυτό ήθελα να πω κύριε Πρόεδρε. Mr. Ευχαριστώ κύριε Μπένιον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τα δικαιώματα που παρέχει η νομοθεσία αυτή σε επιβάτε που αναχωρούν από τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια και που δεν θα συμπεριληφθεί το Γιβραλτάρ εκτό αν συμπεριληφθούν οι τροπολογίε αφορά πολύ βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Η τρέχουσα νομοθεσία δεν ήταν η πιο εύκολη στην υλοποίησή τη. Ειδικότερα όσον αφορά τι εξαιρετικέ περιστάσει. Και η αρχή πολιτική αεροπορία του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα, δυσκολεύεται πολύ με αυτόν τον όρο, το extraordinary circumstances. Ε, βοηθούν λοιπόν οι διευκρινήσει ε, αυτού του όρου. Ελπίζω λοιπόν ότι σήμερα θα δώσουμε σαφήνεια για τις περιπτώσεις τι οποίες μπορεί να λαμβάνει αποζημίωση ε, ένας επιβάτης. Καλωσορίζω επίσης και τις διευκρινήσεις για τις αποσκευές καμπίνας. Και ε, ήθελα να τονίσω και τη δική μου τροπολογία για το άτομο που συνοδεύει κάποιο άτομο με αναπηρία και το δωρεάν εισιτήρια. Θα πρέπει να προσέξουμε για να μην έχουμε περισσότερες ακυρώσεις ε, και αυξημένες τιμές για τους επιβάτες. Ως φιλελεύθεροι δημοκράτες υποστηρίζουμε τα δικαιώματα των επιβατών και πιστεύω ότι αυτό θα παρασχεί ακριβώ αυτή η νομοθεσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, Κομισιό είναι πτήση στα ψηλά για τις εταιρείε, αλλά αναγκαστική προσγείωση για τους επιβάτες. Κύριε Κάλλας, 70% των παραπώνων δεν έχουν καμία ε, απάντηση και επίσης με τον κανόνα των 5 ωρών δεν λαμβάνει υπόψη η απόφαση του δικαστηρίου. Όλα γίνονται υπέρ των αεροπορικών εταιριών. Είναι ακόμα χειρότεροι κανόνες από αυτούς που, τους κανόνες που ίσχυαν που πρόβλεπαν για μια αποζημίωση μετά από δύο ώρες. Στα, στο σιδηρόδρομο μπορεί κανείς με καθυστέρηση μόνο μια ώρας μπορεί να έχει μια ε, αποζημίωση ανεξάρτητα από την απόσταση και αυτό πάντα ισχύει και σήμερα. Αν τελικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι μονάχα να είναι κερδοφόρες οι εταιρείε, κάθε χρόνο παίρνουν 300 δισεκατομμύρια ευρώ ως δώρο από τους Ευρωπαίους φορολογούμενους ενώ οι σιδηρόδρομοι δεν παίρνουν τίποτα και δεν πρέπει να πληρώνουν φόρο για την κυροσύνη καν οι αεροπορικές εταιρείες. Αυτό το μονοπόλιο λοιπόν θα πρέπει να ξεπεράσετε και αυτό είναι δική σας δουλειά. Ευχαριστώ. Κύριε Φλάσακ έχετε το λόγο. Ε, κυρίες και κύριοι η πρόταση για τον ε, κανονισμό περί δικαιωμάτων των επιβατών εξετάζει το ζήτημα από την άποψη των επιβατών και φυσικά πολύ σωστά. Αναφέρομαι στις τιμές, ε, στις ε, πολλαπλές πτήσεις με ανταποκρίσεις σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί η πρώτη πτήση η πληροφόρηση ενημέρωση των επιβατών καθώς και εξαιρετικές περιστάσεις. Καλώς ορίζω όλες αυτές τις διατάξεις. Από την άλλη όμως, ε, παρά τις άριστες προθέσεις, ορισμένα κομμάτια της ε, πρότασης ε, είναι κάπως υπερβολικά φιλοδόξα. Δεν χρειάζεται να διευκολύνουμε τόσο πολύ τα πράγματα για το καταναλωτή. Δεν χρειάζεται οι αερομεταφορείς να χρειαστεί να αυξήσουν τις τιμές τους ώστε να μπορέσουν να τηρήσουν την νομοθεσία αυτή. Πιστεύω ότι χρειάζεται περισσότερο μελέτη το ζήτημα αυτό για να το βελτιώσουμε. Κύριε Πασκόλ. Ντεγκράντε Πασκουάλ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να επενέσω τον εισηγητή. Νομίζω ότι είναι ένα έντονο παράδειγμα τη σημασία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσα στη διαδικασία συναπόφαση και νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προσπάθησε να έχει μια ισορροπημένη πρόταση, λαμβάνοντα υπόψη και τα συμφέροντα των εταιριών και των, και των επιβατών αλλά αυτό ο οποίο θέλει μεγαλύτερη προστασία είναι ο επιβάτης. Αυτό το διορθώνει η έκθεση και υπερασπίζεται το, τα συμφέροντα αυτού του επιβάτη, ο οποίο πολλές φορές είναι τελείω ε, χωρίς καμιά προστασία. Ε, θα ήθελα να επανέλθω λοιπόν σε ορισμένα σημεία, αλλά προηγουμένως θα σας πω ότι οι καθυστερήσεις και οι αποζημιώσεις είναι απαραίτητο να ρυθμιστούν και επίσης η καθυστέρηση στην πίστα απογείωσης που μπορεί να φτάσουν μέχρι τις δύο ώρες είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το τονίσουμε και πρέπει να βρούμε και μια εγγύηση για τις περιπτώσεις πτώχευσης επιχειρήσεων προς όφελος των των επιβατών. Νομίζω ότι όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό ανεξάρτητα από πολιτική παράταξη. Η Επιτροπή Μεταφορών λοιπόν έχει λάβει υπόψη και τη δήλωση του Λονδίνου του 1986 που επιτρέπει να υπάρξει και μία διαδικασία διαλόγου. Μπορούν να έχουν στι χώρες σε περίπτωση διαφωνίας μία άρση των κοινωνικών κανόνων με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μία διαβούλευση μεταξύ τους και έτσι μπορούν να επιληθούν τα προβλήματα. Επομένως αυτό το οποίο έχει λάβει η χώρα ήταν σωστό και επομένως είναι μια σωστή φόρμα. Thank you, Mr. Simpson, Brian. Ο Brian Simpson έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τον συγητή μας και τους σχεδόν συγητέ για την ποιότητα της έκθεσης και επίσης την Κομισιόν, διότι πράγματι αντιμετώπισε το θέμα αυτό. Θα ήταν χρήσιμο να θέσουμε το ερώτημα γιατί γίνεται αυτή η μεταρρύθμιση του κανονισμού 261. Είναι απαραίτητη, κύριε Πρόεδρε, γιατί ο τωρινό κανονισμό έχει τύχει κατάχρηση από τι αεροπορικέ εταιρείε και του βοήθησαν οι εθνικοί ρυθμιστέ σε αυτό το έργο, γιατί ουσιαστικά έχουν αποσύσει κάθε ευθύνη και έχουν με την αδράνειά του ενθαρρύνει τι αεροπορικέ εταιρείε να μπορέσουν να παραβιάσουν την νομοθεσία. Η έκθεση αυτή θέτει τέρμα σε αυτό τον καιρό ευμάρειας και ευτυχίας των αεροπορικών εταιριών. Μόνο 2% των, επιβατών που πλήττονται από καθυστερήσεις ή ακυρίσεις παίρνουν κάποια αποζημίωση. Ένα ισχνότατο και απογοητευτικό 2% γιατί οι εταιρείε λένε ότι όταν υπάρχει κάτι, μια καθυστέρηση, η ακύρωση, όλα αυτά αποσμίωση. σε ανωτέρα βία και προστρέπουν τον κόσμο να αντιμετωπίσει αυτά μόνο στο δικαστήριο. Κλείνει λοιπόν τα παραθυράκια αυτή η έκθεση, τονίζοντας ότι τα τεχνικά προβλήματα δεν αποτελούν λόγο ε, ανωτέρας βίας. Αν χαλάσει το αεροπλάνο σας, λένε στις εταιρείες, δικό σας πρόβλημα είναι αυτό. Επομένως, αν καθυστερήσουν οι επιβάτες ή ακυρωθεί η εταιρεία τους, τότε θα πρέπει να επομιστούν τις ευθύνες τους και να αποζημιώσουν. Κάποιες εταιρείες βέβαια τώρα θα προσπαθήσουν να βρουν νέα παραθυράκια και δεν θα δεχτούν τα δικαιώματα των επιβατών. Αλλά λέω στο Κοινοβούλιο και στους, ε, αεροπορικές εταιρείες ότι αυτή η έκθεση αφορά τα δικαιώματα των ε, επιβατών και όχι τα δικαιώματα των αεροπορικών εταιρείων και πρέπει να υποστηριχθεί από όλους μας. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη Monarch Airlines που μου έδειξε πρακτικά γιατί έπρεπε να κλείσουν τα παραθυράκια. Μετά από μια καθυστέρηση 26 ωρών από την Τενερίφη όταν γύρισα τον Αύγουστο του 2012 η αποζημίωση που δόθηκε στους επιβάτες ήταν τίποτα, ένα μεγάλο τίποτα. Κυρία Μπιλμπά Μπαραντίκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κανονισμός αυτός είναι αναγκαίος για να μπει τάξη σε έναν τομέα προβληματικό όπου συμμετέχουν αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες από διάφορες χώρες και έχει να κάνει με την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Ο ορισμός ε, του κανονισμού αυτού έχει οδηγήσει σε παρεξηγήσεις τώρα. Απλοποιούνται οι διαδικασίες καταγγελίας και εξηγούνται καλύτερα ποιες είναι οι που μπορούν να οδηγήσουν σε αποζημιώσεις. Υπάρχει υποχρέωση καλύτερων υπηρεσιών ε, στα αεροδρόμια ε, προβλέπονται καλύτερες διευκρινήσεις στην πώληση online και εξυπηρετούνται οι χρήστες αεροπορικών εταιριών. Πολύ βασικό αυτό. Πληροφορία, ε, προστασία και βοήθεια. Να υπάρχει κάποιο στο αεροδρόμιο που να μπορεί να εξηγήσει και αποφυγή χρήσεων να μπορεί ο επιβάτης ε, να μπει στο αεροπλάνο ακόμα και αν δεν έχει χρησιμοποιήσει το αλέ του εισιτηρίου του. Έπειτα, ρυθμίστε το θέμα των μουσικών οργάνων στην ε, καμπίνα του αεροσκάφους. Θέματα τα οποία έχουν να κάνουν επίσης με τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή το θέμα της ερμηνείας που οδηγεί σε καταχρήση από ορισμένε αεροπορικές εταιρείε. Ελπίζω να σε γίνουν σεβαστές οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ε, κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δύσκολη δουλειά που έκανε προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των ε, επιβατών, αλλά να φροντίσει και για τη βιωσιμότητα των αεροπορικών εταιριών. Οι επικρίσεις μου έχουν να κάνουν με την αποτυχία που συνοδεύει την τροπολογία για το Γεβραλτάρ. Ποιο είναι το πρόβλημα, ότι δεν υπάρχει δικαιολογία να αποκλείεται το Γιβραλτάρ, οι πολίτε του Γιβραλτάρ που είναι Ευρωπαίοι πολίτε και να μην εφαρμόζονται και σε αυτού τα δικαιώματα επιβατών όπω εφαρμόζονται σε όλου του υπόλοιπου Ευρωπαίου. Πρόκειται για διάκριση που υπονομεύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πού αλλού επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι τέτοιο. Μου φαίνεται πολύ περίεργο που τα μέλη τη Επιτροπή Μεταφορών δεν ε, βοήθησαν να ψηφιστεί η τροπολογία αυτή τη και να σταματήσει η διάκριση αυτή σε βάρο των πολιτών του Γιβραλτάρ. Επίση, θέλω να συμφωνήσω με αυτού που σήμερα καταδικάζουν τη διάκριση αυτή, γιατί οι πολίτε του Γιβραλτάρ αξίζουν περισσότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εμεί γι' αυτό ακριβώ βρισκόμαστε εδώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μαρινέσκο έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Τελευταία έχουμε διαπιστώσει ότι αυξάνονται τα θύματα μεταξύ των επιβατών, θύματα καταχρηστικών πρακτικών από πλευρά των αεροπορικών εταιριών. Σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, οι επιβάτες δεν καταγγέλουν αυτές τις πρακτικές γιατί οι διαδικασίες είναι ιδιαίτερα περίπλοκες ή γιατί απλώ δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Τώρα με την έκθεση αυτή υπάρχει υποχρέωση ενημέρωσης και υπάρχει και υποχρέωση να υπάρχει άτομο επαφή σε κάθε αεροδρόμιο το οποίο θα ενημερώνει τους επιβάτες για τα δικαιώματά του και θα λύνει τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με καθυστερήσει ή ακυρώσει πτήσεων. Έπειτα το θέμα των χειραποσκευών, των αγορών στο αεροδρόμιο. Ε, πρέπει τα πακέτα αυτά, τα αντικείμενα αυτά να μπορούν να μπαίνουν στην καμπίνα του αεροσκάφους επί το όταν υπάρχουν καθυστερήσεις πάνω από δύο ώρες, το ότι οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να προσφέρουν ε, διατροφή και ποτά στους επιβάτες. Το θέμα των αποζημιώσεων επίσης που έχει να κάνει με τις καθυστερήσεις και τις κυρώσεις ενισχύεται με την ρύθμιση αυτή. Επί τα το κατάλογο των απρόβλεπτων καταστάσεων, ώστε να διευκρινίσετε καλύτερα πότε αεροπορικέ εταιρείε πρέπει να δίνουν αποζημιώσεις στου επιβάτε και πότε όχι. Θεωρώ λοιπόν ότι έχουμε πετύχει μια ένα ισορροπημένο κείμενο και ρύθμιση ανάμεσα στα δικαιώματα των επιβατών και τα συμφέροντα των εταιρείων εταιριών και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον συνάδελφο Μπάχα για την τόσο ισορροπημένη έκθεση στην οποία κατέληξε. Ευχαριστούμε κυρία Σενάλοβα Όλγα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα ε, τον εισηγητή μα τον κύριο Μπαχ για την πολυποιωτική του έκθεση. Αποτελεί σημαντικό βήμα προόδου για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών στην αεροπλαγιά. Η τρέχουσα κατάσταση είναι εξαιρετικά σύνθετη. Ως αποτέλεσμα μόνο το 2% των επιβατών οι οποίοι θα μπορούσαν να απαιτήσουν αποζημίωση για καθυστερήσει ακυρώσεις πτήσεων λαμβάνουν ουσιαστικά τέτοια αποζημίωση. Πολύ συχνά οι επιβάτε ε, δεν γνωρίζουν καν τα δικαιώματά του. Γι' αυτό το λόγο χαιρετίζω το γεγονό ε, ότι η έκθεση βελτιώνει σημαντικά την ενημέρωση των επιβατών. ορίζω επίση το γεγονό ότι κατάφερα να περάσω μια τροπολογία στην έκθεση που αφορά τη συμπερίληψη των πληροφοριών για τα δικαιώματα επιβατών στα αεροπορικά ειστήρια. Συγχαίρω τον κύριο Σιγητή για τις ε, διατάξεις που αφορούν τις αποζημιώσεις προς επιβάτες ε, σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας μιας αεροπορικής εταιρείας. Είναι κάτι που προσπαθούμε από το 2009 ε, όταν είχαμε την πτώχευση της Sky Europe και άλλων αεροπορικών εταιρεών εδώ απαιτείται λοιπόν από τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν εξοδικαστικές ε, ε, συμφωνίες ε, για να λαμβάνουν επιβάτες αποζημίωση με τρόπο οικονομικά αποτελεσματικό. Υποστηρίζω λοιπόν την εκτίση. Ευχαριστούμε. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Βότσον. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ την νοτιοδυτική Αγγλία και το Γιβραλτάρ. Αυτό είναι από τα ελάχιστα μέτρα που περιλαμβάνουν για την αεροπλοεία μέτρα τα οποία αποκλείουν το Γιβραλτάρ. Το 2006 η Ισπανία είχε πει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν θα επιδίωκε πλέον την εξαίρεση του Γιβραλτάρ από τέτοια μέτρα για την αεροπλοεία. Πρόσφατα μετέφερε στην Εθνική Νομοθεσία μια νομοθεσία ε, Open Sky που περιλάμβανε το Γιβραλτάρ. Αλλά εδώ παρέμεινε σε αυτή την νομοθεσία η εξαίρεση του Γεβραλτάρ. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Τέθηκε πέρυσι στο Συμβούλιο Μεταφορών και εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών από εμένα και από άλλους. Τόσο στο Κοινοβούλιο όσο και στο Συμβούλιο όλοι αναρωτιούνται γιατί συζητάμε αυτή τη διένεξη εθνικής κυριαρχίας ενώ θα έπρεπε να συζητάμε τα δικαιώματα των επιβατών. Είναι δικαίωμα κάθε Ευρωπαίου πολίτη, είτε είναι από το Γεβραλτάρ, είτε από την Ισπανία, είτε από οπουδήποτε, που χρησιμοποιεί το αεροδρόμιο του Γεβραλτάρ. Προτρύνω λοιπόν του συναδέλφου ε, να ψηφίσουν για τι τροπολογίε 171-174 για να υποστηρίξουμε το λαό του Γεβραλτάρ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Ζήλε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαχ για το δύσκολο εγχείρημα που έφερε σε πέραση με την έκθεση αυτή και να τονίσω ορισμένες από τις βασικές αρχές που διέπουν αυτή την απόφαση. Από εδώ και πέρα οι αεροπορικές εταιρείες δεν θα είναι σε θέση να ακυρώνουν πτήσεις επιστροφής μόνο και μόνο γιατί κάποιος δεν χρησιμοποίησε την πτήση ΑΛΕ. Ακυρώνει το ειστήριο δηλαδή. Είναι σαν να έχετε μία συνδρομή για μία σειρά από παραστάσεις στην όπερα στο θέατρο και άμα δεν, δεν παραστείτε σε μία παράσταση χάνετε τις υπόλοιπες. Υπάρχουν ορισμένες επίσης φθηνές αεροπορικές εταιρείες που κρατούν τους επιβάτες τους για ώρες στα αεροδρόμια μέσα στο αεροπλάνο, στην πίστα, λόγω καθυστέρησης και αυτό θα καταργηθεί. Και επίσης η έκταση περιστάσεις δεν θα είναι πια ε, καταχρηστικές. Ο κύριος Πίρκερ, κύριε πρόεδρε, οι ρυθμίσεις προς όφελος των εκατομμυρίων επιβατών που πετούν στην Ευρώπη κάθε μέρα είναι πάρα πολύ σημαντικές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαίρομαι για το γεγονός ότι υπάρχει μια σειρά από πολύ καλές λύσεις οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν και ελπίζω θα εγκριθούν αύριο που θα συμβάλλουν στην βελτίωση την ουσιαστική βελτίωση της πρότασης Κομισιόν. Είναι, η, είναι ο εισηγητής ο οποίος το έχει επιτύχει αυτό. Απλώς θέλω να σταθώ όμως σε ορισμένα σημεία. Πρώτα απ' όλα έχουμε πετύχει οι αποζημιώσεις για περίπτωση καθυστέρησης να γίνουν πιο απλές και να αυξηθούν. Επίσης, ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια πολιτική no-show όταν κανείς δεν έχει πετάξει το πρώτο κομμάτι μιας πτήσης με επιστροφή, διατηρεί την, ε, την ε, επιστροφή. Επίσης τα θέματα των τεχνικών προβλημάτων. Υπάρχει ένας σαφέστερος ορισμός ο οποίος θα ισχύει και δεν μπορούν επομένως οι εταιρείε να χρησιμοποιούν αυτό το κόλπο και το ίδιο ισχύει και για τις χειραποσκευές. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι η δημιουργία των σημείων πληροφόρησης και παραπώνων ώστε να μην μπορούν οι εταιρείες να αρνούνται να παρέχουν πληροφορίες. Είναι απαραίτητο επίσης σε περίπτωση παραπώνων να υπάρχει ταχεία αντιμετώπιση. Και χαίρομαι λοιπόν που υπάρχουν αυτές οι λύσεις υπέρ των ε, επιβατών. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Λάιχτφριντ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να σας συγχαρώ κύριε Σιγητά γιατί είναι μια πολύ καλή έκθεση και χρειάστηκε σκληρή δουλειά γιατί ήταν σαφές από την αρχή ότι υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να βελτιωθούν στην φιλική προς αεροπορικές εταιρείες της Επιτροπής. Δεν ήταν μια πρόταση υπέρ των επιβατών, αλλά υπέρ της κερδοφορίας των αεροπορικών εταιρών. Έχουν γίνει λοιπόν σημαντικές βελτιώσεις, ιδίως σε ό,τι αφορά τις χειραποσκευές και επίσης σε ό,τι αφορά θέματα εκτάκτων περιστάσεων έχουμε εξασφαλίσει λοιπόν να υπάρχει καλύτερη ουσιαστική αρρωγή προς τους επιβάτες οι οποίοι βρίσκονται σε ένα αεροδρόμιο και δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Με την πρόταση αυτή λοιπόν έχει εξασφαλιστεί καλύτερη προστασία των επιβατών και έχει δημιουργηθεί και ένα σύστημα το οποίο εμποδίζει τις αεροπορικές εταιρείες όταν σε πολλαπλές πτήσεις χάνει κανείς μια πτήση να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει τις υπόλοιπες. Δεν υπάρχει κάποιος αποχρόν λόγος για κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται, δεν είχε νόημα ο επιβάτης να πρέπει να ξαναπληρώνει για μια πτήση που είχε ήδη πάρει. Είναι θετικό λοιπόν ότι το Κοινοβούλιο έχει τροποποιήσει την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όφελος των καταναλωτών, προς όφελος των εκλογέων μας και εν των επικειμένων ευρωπαϊκών εκλογών. Είναι καλό να ξέρουν οι πολίτες ότι δεν σκεφτόμαστε μόνο τη βιομηχανία αλλά και τους ανθρώπους. Ο κύριος Higgins. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όπως και προλαλήσατε, έτσι και εγώ θέλω να συγχαρώ τον φίλο και συνάδελφο Τζόρτζο Μπαχα για το εξαίρετο έργο του για αυτή την έκθεση. Όπως γνωρίζουμε, Πρόεδρε, ο κλάδος έχει περάσει από πολλές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Έχουν αυξηθεί οι επιβάτες και υπάρχει και ελευθέρωση στην αγορά. Καλό αυτό βέβαια για χώρες όπως και η Ιρλανδία που εξαρτάται πολύ από τις αερομεταφορές. γι' αυτό χρειάστηκε κατάλληλη όμως ρύθμιση αθέμητος ανταγωνισμός κατά χρηστικές εμπορικές πρακτικές είναι κάτι το οποίο δεν θέλουμε. Από τότε που άρχισε να ισχύει ο κανονισμός το 2004 υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τις διαφορετικές ερμηνείες που οδηγούν σε γκρίζες ζώνες και παρεξηγήσεις. Οι επιβάτες δυσκολεύονται πρώτα απ' όλα να απαιτήσουν τα... τη δικαίωσή τους και από την άλλη μεριά δεν γνωρίζουν καλά καλά ποια είναι τα δικαιώματά τους γιατί οι αεροπορικές εταιρείε δεν τους ενημερώνουν σχετικά. Το κοινοβούλιο μας λοιπόν έχει ήδη εκφράσει την άποψή του και παλιότερα για τα θέματα αυτά με διάφορα ψηφίσματα το 2012. Γι' αυτό λοιπόν κύριε Πρόεδρε χαίρομαι πολύ που τώρα έχουμε σαφήνεια όσον αφορά τις αποζημιώσεις, όσον αφορά τις καταγγελίες, όσον αφορά την ε, ενημέρωση και το, το κόστος. Όλα αυτά θα βοηθήσουν και τα μικρά αεροδρόμια να συνεχίσουν να αναπτύσσονται και να μεγαλώνουν και θα βοηθήσει διάφορες περιφέρειες μεταξύ των οποίων και αυτή που εκπροσωπώ εγώ εδώ. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σφίτσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Οι πολίτες μου πολλές φορές με ρωτάνε επειδή είμαστε νέα χώρα μέλος τι κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μας. Τι κάνετε για μας. Νομίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή είναι ένα καλό παράδειγμα για να τους εξηγήσω τι κάνουμε. Είμαι από την Κροατία όπως γνωρίζετε και το 5% του ΕΠΑΣ έρχεται από τον τουρισμό. Οι αερομεταφορές είναι κάτι πολύ σημαντικό για τον τουρισμό. Εγώ έρχομαι από το Ντουμπρόβνικ και εμείς εξαρτώμαστε πάρα πολύ από τους τουρίστες που έρχονται αεροπορικώς στη χώρα μου. Πολύ σημαντικό θέμα λοιπόν αυτό για μένα και πολύ σημαντικό που μπορώ να διαπιστώσω ότι πια οι επιβάτες μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις, να επιβάλλονται τα δικαιώματά τους που υπάρχουν συγκεκριμένα όρια και νομίζω ότι Όλα τα δικαιώματα τα οποία προτείνει στην έκθεσή του ο κύριο Βαχ πρέπει να επιβληθούν. Τον συγχαίρω λοιπόν γιατί νομίζω ότι έκανε πολύ καλή δουλειά και ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε προ την ίδια κατεύθυνση να βελτιώνουμε τα δικαιώματα των επιβατών όχι μόνο τις παραμονές των ευρωεκλογών, αλλά θα συνεχίσουμε να έχουμε υπόψη μας τα δικαιώματά τους και μετά. Όλοι αυτοί οι κανόνες πρέπει να εφαρμόζονται με τον ίδιο τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση όταν πρόκειται για τους καταναλωτές. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κόζα τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Μπαχ έχει επιτελέσει εξαίρετο έργο όλα αυτά τα χρόνια σε σχέση με τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών εταιριών. Θυμάμαι πριν από μερικά χρόνια συζητούσαμε για το δικαίωμα των ε, επιβατών και ήταν πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβω πώς είναι δυνατόν άτομα με αναπηρίες, άτομα με αναπηρικές καρέκλες ή άλλες ε, δυσκολίες δεν μπορούσαν να βρίσκονται στην ίδια θέση όπως και οι υπόλοιποι. Χαίρομαι λοιπόν που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τώρα το αντιλαμβάνεται αυτό, σε αντίθεση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό που με την πρόταση του Βαϊκού Κοινοβουλίου διορθώθηκε αυτό. Χαίρομαι επίσης για την μεγάλη πρόοδο ε, γενικά για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Οι αεροπορικές εταιρείε και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας. Πρέπει να προσφέρουν ένα σύστημα με διαφάνεια όσον αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα. Χαίρομαι επίσης που συμμετείχαν και μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες οργανώσεις και χαίρομαι επίσης που η νομοθεσία πια απαιτεί και προσωπική εξυπηρέτηση, γιατί αυτό σημαίνει ισότητα στην πραγματικότητα. Ο κύριος Ανδρέας Σουάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θέλω να συγχαρώ την Κομισιόν για το γεγονός ότι είχε την πρωτοβουλία να υποβάλει αυτή την πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χωρίς αυτή την πρόταση τα δικαιώματα των επιβατών δεν θα μπορούσαν να προωθηθούν. Βέβαια το γεγονός ότι υπάρχει βελτίωση, υπάρχουν δυνατότητες βελτίωση στην πρόταση τη Κομισιόν και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο. Το βασικό πρόβλημα για του επιβάτε δεν είναι το θέμα της παροχής αποζημίωσης. Το θέμα είναι όταν έχουν προγραμματίσει να πάνε κάπου να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους εγκαίρως. Αυτό είναι το βασικό. Η ακρίβεια στις πτήσεις. Και δεν πρέπει να θέσουμε εμπόδια με τις αποζημιώσεις. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είναι προβλέψιμη η άφηξη των επιβατών εκεί που θέλουν να φτάσουν. Και γι' αυτό είναι απαραίτητο να υπάρξει ένα σύνολο κανόνων που να είναι λειτουργικός. Αυτό ελέγχθη σήμερα ότι έχουμε εξασφαλίσει μια πρόοδο, αλλά στην περίπτωση που, υπάρχει πολλές φορές μια καθυστέρηση, οι αεροπορικές εταιρείες επικαλούνται ανωτέρα βία ή τεχνικά προβλήματα. Και χαίρομαι κύριε Επίτροπε, αν μπορείτε να εξασφαλίσετε ότι πράγματι θα τηρήσουν αυτό τον κανόνα οι αεροπορικές ή θα δυσκολέψουν ή θα δυσκολέψουν την εφαρμογή των δικαιωμάτων των επιβατών. Ευχαριστώ. Έρχομαστε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω τη δυνατότητα να δώσω πέντε, το λόγο σε πέντε συναδέλφους, ξεκινώντας με τον κύριο Μπάνκι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είμαι ευγνώμων προς τον κύριο Μπαχ για αυτή την πολύ σημαντική έκθεση που εκπώνησε. Κάθε χρόνο η αεροπορία και η, κίνηση, η αεροπορική κίνηση επεκτείνεται και αυτό θα συνεχιστεί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να διασφαλίσουμε την ασφάλεια και την άνεση των επιβατών καθώς και τη ε, μη καθυστέρηση των πτήσεων. Είναι σημαντικό λοιπόν να ρυθμίσουμε τη, σωστά τις αποζημιώσεις προς τους επιβάτες ώστε οι αερομεταφορείς ε, να παίρνουν στα σοβαρά αυτή τους την υποχρέωση. Η νομοθεσία αναφέρει επίσης ότι πρέπει να δημιουργηθούν σημεία επαφής, ε, σημεία επαφής όπου θα μπορούν να απαιτήσουν την αποζημίωση τους επιβάτες και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πέτραγκας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεδομένη συμπεριφορά ορισμένων αερομεταφορέων που μου λένε πολύ ψηφοφόροι μου στην Ιρλανδία, αυτή η αναθεώρηση τη νομοθεσία για τα δικαιώματα των επιβατών είναι ιδιαίτερα επίκαιρη. Πολύ συχνά οι αερομεταφόροι δεν παρέχουν την αρρωγή στου επιβάτε που έχουν δεσμευτεί μέσω τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία να προσφέρουν εκμεταλλεύονται την άγνοια των επιβατών ε, και τα νομικά παραθυράκια. Πολλές υποθέσεις που ε, ε, εμφανίζονται μπροστά στα δικαστήρια δείχνουν ότι χρειάζεται να διευκρινιστούν οι κανόνες για όλα αυτά. Η αποζημίωση για τις καθυστερήσεις εισάγονται και βάσει τη αποφάσης του δικαστηρίου. Ε, αναμένω προσδοκώ το δω την εφαρμογή της ε, νομοθεσίας αυτής και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε κύριος Νικολάσιτς. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, η αγορά αεροπορικών μεταφορών έχει απορριθμιστεί είναι καλύτερο μερικές φορές για τους επιβάτες. Από την άλλη μεριά όμως έχει χαλάσει ποιότητα. Και κάποιες αεροπορικές εταιρείες προχωρούν σε αθέμητο ανταγωνισμό σε βάρος των επιβατών. Υπάρχουν νομικά κενά τα οποία επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να μην φέρουν σε πέρας τις υποχρώσεις τους. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο να μην μπορούν οι επιβάτες να παίρνουν την πτήση τους επειδή προηγουμένως δεν χρησιμοποίησαν το προηγούμενο κομμάτι του εισιτηρίου τους. Έπειτα, χαίρομαι που τώρα προβλέπεται οι αεροπορικές εταιρείες να ενημερώνουν έγκαιρα τους επιβάτες για τα δικαιώματά τους. Ε, χαίρομαι επίσης για το ότι υπάρχει έντυπο ενιαίο καταγγελιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλες τις γλώσσες. Ευχαριστούμε. Κύριος Στανέλης. Η μεταρρύθμιση του ισχύοντος κανονισμού είναι αναγκαία ώστε να κλείσουμε τα κενά που γνωρίζουμε πως υπάρχουν και κυρίως να τον εφαρμόσουμε πλήρως. Η μεταρρύθμιση αυτή πρέπει να υπερασπιστεί την εφαρμογή του κανονισμού στην οποία εστιάζονται και τα περισσότερα προβλήματα ένα ελάχιστο μόνο ποσοστό των επιβατών που δικαιούνται αποζημίωση τη λαμβάνουν και αυτό μάλιστα μετά από μαραθώνιες προσπάθειες. γι' αυτό τον λόγο από την πλευρά των σοσιαλιστών ενσωματώσαμε στο κείμενο νέα μέτρα που έχουν στόχο την ενδυνάμωση αυτής της διάστασης. επίσης σημαντική για τους επιβάτες θα είναι η θεσμοθέτηση του αυτονόητου δικαιώματος μεταφοράς των αγορών τους από το αεροδρόμιο καθώς επίσης και το ξεκαθάρισμα του ζητήματος της μίας χειραποσκευής που καταχρηστικά εφαρμόζεται από όλο και περισσότερες αερομεταφορείς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Τικάου. Έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αγαπητέ κύριε Συγητά, θα ήθελα να συγχαρώ ιδιαίτερα τον Συγητή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά τα δικαιώματα των ε, επιβατών, ιδίω για την παροχή πληροφορία και αρρωγή. Οι εθνικέ αρχέ θα πρέπει επίση να εφαρμόσουν πρόστιμα σε αεροπορικέ εταιρείε που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ενάντια των επιβατών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για του επιβάτε να έχουν σαφή νομοθεσία η οποία καλύπτει τα δικαιώματά Του Πρέπει να εξασφαλίσουμε και ότι δεν θα υπάρχουν παραθυράκια που επιτρέπουν σε αεροπορικέ εταιρείε να εκμεταλλεύονται την νομοθεσία σε βάρος των επιβατών. Θέλω να υπογραμμίσω τις σημαντικές βελτιώσεις που έχουν επέλθει για την παροχή πληροφοριών σημεία παραπώνων στα αεροδρόμια, την απλοποίηση των διαδικασιών για την υποβολή παραπώνων, τους απλοποιημένους κανόνες για τις βαλίτσες και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχει Έχουμε ακόμα τρία άτομα που ζήτησε, ζήτησαν το λόγο στη διαδικασία Καστιά. Κυρία Όμεν Ρόιτεν πρώτα. Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ και εγώ τον συνάδελφο Μπάχα για το εξαίρετο αποτέλεσμα στο οποίο κατέληξε. Χαίρομαι επίση πολύ που οι τροπολογίε του κυρίου Μπάχα έχουν συμπεριληφθεί και που δίνουμε πια ιδιαίτερη σημασία στις διαφορετικέ ερμηνείε. Όντως ο χειρισμός πρέπει να γίνεται καλύτερα από ό,τι στον αρχικό κανονισμό και να επωφελείται το κοινό. Ο καταναλωτής δεν πρέπει να ανακάζεται να πηγαίνει στο δικαστή, χαίρομαι που προβλέπονται και εξοδικαστικές ε, διαδικασίες. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να μπορεί φτηνά να καταφεύγει στη δικαιοσύνη εφόσον χρειαστεί ο καταναλωτής και να γνωρίζει τις διαδικασίες. Στην ε, Ολλανδία δυστυχώς δεν υπάρχει ισορροπία και ίδιες συνθήκες για όλους εξαρτάται από το ποια εταιρεία ανήκει σε ποιο όργανο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να διορθωθεί ελπίζω στο Συμβουλίο. Κυρία Κάντεμαχ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε και εγώ χαιρετώ τις ε, προσπάθειες του κυρίου Μπάκ και τις πολλές τροπολογίες που κατέθεσε. Θα ήθελα όμως να εξάρω δύο σημεία. Το ένα είναι ότι υπάρχει στο μέλλον δυνατότητα οι άνθρωποι με προβλήματα κινητικότητας να πετούν πιο εύκολα και επίση το να ληφθεί υπόψη το δικαίωμα των επιβατών σε περίπτωση καθυστερήσεω ή ακύρωση πτήση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση να υπάρχουν σαφεί συνομιλητέ οι οποίοι πρέπει να δώσουν ακριβεί πληροφορίε σε σχέση με τι πτήσει. Έχουμε ζήσει την εμπειρία αυτή με το σύννεφο τέφρας όταν οι επιβάτε δεν μπορούσαν να έχουν καμιά πληροφορία και ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα, ιδίω για του πιο ηλικιωμένου επιβάτε, οι οποίοι δεν είχαν καμία πρόσβαση στο διαδίκτυο να ξέρουν τι θα γίνει και να έχουν κάποια πληροφόρηση σε σχέση και με, την, με τα δικαιώματά του και για αυτού οι οποίοι πρέπει να στεγάζονται για να διανυκτερεύσουν λόγω μια καθυστέρηση, νομίζω ότι έχει επέλθει μια σημαντική βελτίωση επίση. Η κυρία Μόζερ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ περίεργο που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα, διότι υπάρχουν καλοί κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα των επιβατών όσον αφορά ακυρώσεις και καθυστερήσεις. Το πρόβλημα είναι ότι οι αερομεταφερείς δεν τηρούν τους κανόνες αυτούς. Καλό είναι λοιπόν που η Κομισιόν αποφάσισε να καταστήσει πιο σαφείς τους κανόνες αυτούς. Ωστόσο, δεν είναι καλό που έγιναν πολύ αυστηροί αυτοί οι κανονισμοί. Προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε όλα αυτά, αλλά κατά την άποψή μου δεν ε, έχουμε πάει αρκετά μακριά. Πρέπει να προστατέψουμε τους επιβάτες. Μιλάμε για απρόβλεπτες καταστάσεις όπως μια απεργία. Γιατί απεργία είναι απρόβλεπτη κατάσταση γιατί δεν μεταχειρίζονται απλά σωστά το προσωπικό του, ώστε να μην κατεβαίνει σε απεργία και αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε προστασία τόσο του προσωπικού όσο και των επιβατών και δεν θα βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει τη διαδικασία. Καστία, δεν το λόγο στον κύριο Κάλλας. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση, για το έργο το οποίο επιτελέσατε και σίγουρα θα συνεχίσουμε τις επικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων. Το επόμενο βήμα είναι, ελπίζει η Επιτροπή, ότι το Συμβούλιο θα μπορέσει να καθορίσει τη δικιά του θέση όσον αφορά αυτή τη τόσο σημαντική νομοθετική πρόταση και ότι έτσι θα μπορέσουν γρήγορα να, μετά τις εκλογές να αρχίσουν οι διοργανικές συνομιλίες. Η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ότι η αναθεώρηση του κανονισμού αυτού αποτελεί σημαντική βελτίωση για τους επιβάτες. Γιατί τώρα πια έχουμε πιο σαφείς, πιο συγκεκριμένους, πιο καλά εφαρμόσιμους ε, κανόνες και ρυθμίσεις όσον αφορά την, ε, τις αεροπορικές μεταφορές. Επίσης προσπαθήσαμε να βρούμε και μια ισορροπία ανάμεσα στα δικαιώματα των επιβατών και τα συμφέροντα των αεροπορικών εταιριών γιατί και οι αερομεταφορείς λειτουργούν μέσα σε δύσκολες συνθήκες σήμερα και στο κάτω-κάτω δεν είναι οι εχθροί των επιβατών, θέλουν να μεταφέρουν επιβάτες και να κερδίσουν βέβαια έσοδα από την μεταφορά αυτή. Άρα πρέπει να υπάρχει μια καλή ισορροπία. Πιστεύω ότι αυτό που καταφέραμε να αποφύγουμε είναι τις ακυρώσεις πτήσεων, που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί και για τους επιβάτες και για τους αερομεταφορείς. Συνεπώς, για να πηγαίνουν οι επιβάτες στον προορισμό τους, όποιος και αν είναι αυτός, αυτή ήταν η κύρια προτεραιότητά μας κατά την εκπόνηση της πρότασής μας και κατά την συζήτηση εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Τελευταίος αλλά όχι ίστατος ο κύριος Μπάχο εισηγητής. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και προφανώς ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για την ευρεία υποστήριξη που μου έδωσαν. Ο στόχος μας ήταν πραγματικά να είμαστε φιλόδοξοι και να έχουμε μια θαραλέα έκθεση. Αυτό το πετύχαμε. Και πραγματικά απογοητεύομαι για το Συμβούλιο δεν έχει δείξει την κατάλληλη φιλοδοξία. Ελπίζω, κύριε Κάλλας, ότι θα πιέσετε το Συμβούλιο να προωθήσει το θέμα αυτό προς το συμφέρον των επιβατών. Υπάρχουν ορισμένε αεροπορικέ εταιρείε που από ό,τι ξέρω έχουν ήδη απαντήσει στην αίτησή μα. Έχουν θεσπίσει νέου κανόνε για τι χειραποσκευές και αυτό το χαιρετίζω ω μια θετική εξέλιξη. Είχε πολλέ προτάσει η συζήτηση, θα ήθελα να σταθώ μόναχα με ορισμένα σημεία το υψηλό κόστος για τις επιχειρήσεις από τις διαμαρτυρίες μα μόνο, και τις αποζημιώσεις. Μα μόνο 2% των ε, επιβατών έχουν ε, πάρει αποζημιώσεις και οι αποζημιώσεις αυτές δεν εμφανίζονται με ε, εμφανή τρόπο στους ισολογισμούς των εταιριών. Έχω εκφράσει τις ανησυχίες μου ότι δεν μπορεί να δυσκολευτεί η δυνατότητα διεκδίκησης των αποζημιώσεων στα δικαστήρια από τους επιβάτε. Επίσης για τα μουσικά όργανα στον θάλαμο επιβατών. Το έχουμε ρυθμίσει το θέμα αυτό. Και επίσης για το θέμα ανα, ε, αλλαγής ε, της διαδρομής. Και εκεί έχουμε ένα θετικό βήμα προς όφελος των επιβατών. Ο κανόνας των τριών ε, ορών που μπορεί να οδηγήσει σε ακυρώσει πτήσεων. Εγώ νομίζω ότι η φόβη αυτή είναι αβάσιμη. Νομίζω ότι οι αεροπορικέ εταιρείε έχουν τη δυνατότητα να οργανωθούν σωστά για να αντιμετωπίσουν μικρά προβλήματα αυτού του είδου. και επομένω, μέσα σε τρει ώρε, αν δεν είναι ένα μείζον πρόβλημα μπορούν να εξασφαλίσουν τα φύγη φύγει η πτήση. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την υποστήριξή σα και ελπίζω ότι θα έχουμε θετική απόλυξη αύριο. Ευχαριστώ. Τον κύριο Μπάχ έχει τελειώσει η συζήτηση. Αύριο η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 12. Ερχόμαστε στο επόμενο σημείο που είναι η έκθεση Μωράες για τους εποχιακούς εργαζόμενους από τρίτες χώρες. Και θέλω να δώσω τώρα τον λόγο στον εισηγητή.